παράγραφος 2 του κανονισμού. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εισηγητές να παρουσιάζουν τις εκθέσεις εντάχει. Ξεκινώ με την έκθεση του κυρίου Μπέλντερ. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάλια. Για τέσσερα λεπτά δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλντερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα κάνω την παρουσίαση αυτή της έκθεσής μου για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίες και κύριοι δεν μπορεί πλέον ε, να συνεχίσει δεν υπάρχει δεν μπορεί πια να συνεχίσει απλώς να δίνει τις υποσχέσεις που έδωσε στη Θεσσαλονίκη το 2003 στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Κάποια στιγμή τα λόγια θα πρέπει να γίνουν και οι ρητορικοί θα πρέπει να γίνουν πράξεις. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρή ευθύνη σχετικά και ο, θυμίζω την Σρεμπερνίτσα και τη σχετική συζήτηση ε, με άλλα λόγια η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξεκινώ ε, λέγοντας ότι θα πρέπει να κάνουμε να εφαρμόσουμε, να ξεκινήσουμε ένα σύμφωνο σταθερό ένα μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ε, με τις χώρες αυτές πράγμα το οποίο θα τις βοηθήσει ιδιαίτερα προετοιμαστούν για την, ε, ε, το ευρωπαϊκό τους μέλλον αν θέλετε για την ένταξή τους προσπάθησα όταν ξεκίνησα την έκθεση αυτή να δω ποια είναι η κατάσταση. Πήγα στη Χάγη, στο δικό μου ε, Υπουργείο Οικονομικών για να δω πώς έχουν τα πράγματα και πραγματικά μεγάλη μου χαρά είδα ότι η Ολλανδική τουλάχιστον κυβέρνηση δέχεται ε, να έρθει σε επαφή με τις ε, κυβερνήσεις των χωρών αυτών για να δουν ακριβώς τι που μπορούν να βοηθήσουν και ποια είναι τα πραγματικά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ε, το βάζω αυτό στην έκθεσή μου όχι επειδή είναι Ολλανδικό παράδειγμα αλλά επειδή πιστεύω ότι η μέθοδος αυτή αποδίδει καρπούς και είναι καλύτερη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. επόμενο θέμα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η ενεργειακή πολιτική. Θα είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ε, έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή αυτή για την ε, ανάγκη θέσπισης μιας κοινή ε, ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε ποια είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και πώς ορισμένοι μπορούν πολύ εύκολα να αφήσουν στην παγωνιά ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης τότε δεν χρειάζεται ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται υπό αυτές τις συνθήκες να ξανατονίσω πόσο αναγκαία είναι μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε όλοι μαζί, μαζί και με την Επιτροπή Διεθνούς ε, Εμπορίου να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς ε, κάναμε ε, κάποια ταξίδια στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων ήδη. Ε, δεν πήγαμε σε όλα τα μέρη που θα θέλαμε να είχαμε πάει βεβαίως, αλλά, αλλά νομίζω ότι μέσω μιας ενεργητικής, ενεργειακής πολιτικής πραγματικά ή μια κάποιων σχετικών συζητήσεων θα φέρναμε τις χώρες αυτές κοντύτερα στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πραγματικά θεωρώ ότι η έκθεση μου αυτή είναι ένα πρώτο βήμα στο επόμενο βήμα θα πάμε στην καθεμία χώρα χωριστά η Κυρία Βασιλείου να σας συγχαρώ καταρχάς ε, και βουλευτά η έκθεση σας έχετε σε μια χρονική στιγμή που τα Δυτικά Βαλκάνια προσεγγίζουν όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει μια συνολική εικόνα των θεμάτων που διακυβεύονται στις εμπορικές, οικονομικές και, και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δυτικών Βαλκανίων και Ευρώπης. Ναι. Θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα στην έκθεσή σας. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι αξιόλογος και πολύτιμος ε, εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάρτιο του 8 η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια επαναλαμβάνει την δέσμευση της Ένωσης εν ώψη της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου της Κεντρικής Ευρώπης για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η Επιτροπή συμφωνεί με τον εισηγητή ότι η προοπτική προσχώρηση στην Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για την εξασφάλιση της ειρήνης και της αφαιρότητας στην περιοχή. Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης ότι η τήρηση και η εκπλήρωση από κάθε κράτος μέλος των κριτηρίων της Κοπενχάγης είναι εξαιρετικά σημαντική όταν εξετάζουμε την ετοιμότητα προσχώρησης μιας χώρας στην Ένωση. Η Ένωση είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος των Δυτικών Βαλκανίων. Βαθύτερες ε, οικονομικές, ε, βαθύτερη οικονομική δεσμή λοιπόν μεταξύ Βαλκανίων και Ένωσης είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της περιοχής. Όπως τονίζεται σωστά στην έκθεση, η απελευθέρωση του εμπορίου και η ε, οικονομική ενοποίηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ε, διαδικασία σύνδεσης και εμείς βοηθήσαμε στο πλαίσιο αυτό τα Δυτικά Βαλκάνια σε τρία επίπεδα. Πρώτον, σε διμερές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια ήδη από το 2000 για να διευκολύνει την πρόσβαση των εξαγωγών της, ε, προς, των εξαγωγών της περιοχής στις αγορές της Ένωσης. Ε, διαπραγματευθήκαμε τρεις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών σε τμήμα των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης για να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να διευρύνουμε και να διευκολύνουμε την προσχώρηση, την ευθυγράμμιση των χωρών ε, των Βαλκανίων με την Ένωση, κυρίως στο επίπεδο του κοινωνικού, του κοινωνικού εκτιμένου. Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο διευκολύναμε τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης και αποφασίσαμε να παράσχουμε οικονομική βοήθεια και τεχνική βοήθεια στην γραμματεία της ε, ε, δομής αυτής και να βοηθήσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντική σημαντικό το γεγονό ότι η συμφωνία θα θεωρείται ίδιον της περιοχής και θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την ενδοπεριφερειακή ένταξη και εν ώψη της πλήρους συμμετοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, η ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δημιουργεί τις υποδομές για να συζητήσουμε εμπορικά θέματα και σε περιφερειακό και σε διμερές επίπεδο. Κάτι ουσιαστικό για να διευκολύνουμε και να ε, εμβαθύνουμε την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της ε, συμφωνίας και θα συνεχίσει να ε, παρουσιάζει τις εξελίξεις στην ετήσια έκθεση που παρουσιάζει κάθε χρόνο για την ενταξιακή και προενταξιακή διαδικασία των χρόνων αυτών. Τρίτον, σε πολυμερές, σε, πολυ, σε πολυμερές επίπεδο, εμείς υποστηρίσαμε την προσχώρηση των χωρών της περιοχής στον ΠΟΕ, καθότι κάτι τέτοιο είναι βασικό αναγκαίο βήμα για την πραγματική και αποτελεσματική συμμετοχή των χωρών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε όλα τα εργαλεία πολιτικής που διαθέτει για να υποστηρίξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στις προσπάθειές τους να να μεταρρυθμιστούν και να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο. Τα εργαλεία προενταξιακή επικουρία είναι σημαντικά για να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμε ανάγκε ανάπτυξη των χωρών. Η συμμονολική χρηματοδότηση του παρόντο δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 ανέρχεται σε 11,5 δις ευρώ. 11,5 δις. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με όλες τις εμπλεκόμενες της περιοχής χώρες για να δημιουργήσει οδικούς χάρτης για την άρση των καθεστώτων θεώρησης. Θέλω επίσης να σας, να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις και να φέρει τις οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων όσο εγκύτερα γίνεται στις οικονομίες της Ένωσης. Θέλω Εν τέλει, να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεσή του και με χαρά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται την γενική του προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Και τώρα η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί αύριο. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της κυρίας Μαγκίνης που έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε και πρόεδρε κύριε Επίτροπε,